θετικές ε, αλλαγές ε, οι οποίες θα προετοιμάσουν ένα σωστό μέλλον θα συνεχίσουμε και τη στρατηγική μας έτσι όπως την ε, έχουμε εκπονήσει μέχρι τώρα. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Άστον, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής ε, και είπα τη εκπρόσωπε. Ακούσαμε με προσοχή τα όσα μας είπατε για την Κυργυζία. Τώρα θα, ακούσουμε, θα σας ακούσουμε την ίδια προσοχή να μας μιλάτε για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Ε, να σας πω ότι... Έχω δεχθεί τρεις προτάσεις ψηφίσματος ή μάλλον όχι διορθώνει ο Πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτό. Πρόκειται για ανακοίνωση η οποία θα ε, αναγνωστεί μετά το πέρας της συζητήσεως και επομένως δίνω αμέσως τον λόγο στην ε, ε, Λέδη Άστον έτσι ώστε να κάνει την εισήγησή της όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Ο Καναδάς περας της συζητησεως και επομένω δινω αμεσως τον λογο στην λεδη αστον ετσι ωστε να κανει την εισηγηση τη οσον αφορα τη συνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση καναδα ο καναδας βεβαιως ειναι ένας από τους παλαιότερους και κοντινότερους εταίρους της Ένωσης. Συνεργαζόμαστε σε πολλά ζητήματα, διμερεί και παγκοσμίω. Η σχέση μας βασίζεται στην κοινή μας ιστορία που είναι βεβαίως μακροχρόνια και έχουμε και κοινέ αξίες και οπότε πρέπει να προστατεύσουμε και τα κοινά μας συμφέροντα και για το συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης και του Καναδά αλλά και για την ασφάλεια την παγκόσμια. Οπότε είναι μια σημαντική σχέση. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν για να μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρω. Και αυτό είναι ο στόχο τη επόμενη Συνόδου Κορυφή που θα λάβει χώρα στι Βρυξέλλε 5 Μαου. Η συγκυρία είναι ευτυχή γιατί σημαίνει πως ο Καναδάς προεδρεύει στη συνόδους G8 και G20 και μπορούμε άρα να κάνουμε έναν απολογισμό και να δούμε ποια ζητήματα θα μας απασχολησουν συνοδος συνόδους G8 και G20, π.χ. πώς θα έχουμε μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, ρύθμιση των χρηματαγορών, κλιματική αλλαγή και μη διάδοση των πυρηνικών όπλων ήμουν πρόσφατα στην συνεδρία των G8 στον Καναδά που συζητήθηκαν πολλά από αυτά τα ζητήματα. Επίσης θα συζητήσουμε τις διμερείς σχέσεις και το πώς θα συνεργαστούμε σε περιφερειακές κρίσης. Στόχος μας είναι να έχουμε μια σοβαρή συνάντηση. Θα δούμε λοιπόν το πώς θα εξυγχρονιστεί η διμερής μας σχέση, το πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο μια φιλόδοξη εμπορική και οικονομική συμφωνία. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση της προόδου από την τελευταία σειρά διαπραγματεύσεων, αλλά θα δοθεί και νέα ορμή στις διαπραγματεύσεις ε, λαμβανομένης υπόψη τη σημασία τους για το εμπόριο και τις θέσεις εργασίας. Για το εμπόριο θα στείλουμε το μήνυμα πως είμαστε και οι δύο κατά του προστατευτισμού και θα επαναβεβαιώσουμε την δέσμευσή μας για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στον γύρο της Ντόχα. Επίσης θα επιβεβαιώσουμε την δέσμευσή μας για αμοιβαία απαλλαγή από βίζα για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα δούμε την συνεργασία μας στην αντιμετώπιση κρίσεων. Έχουμε πάρα πολλές συνεργασίες, π.χ. στην αστυνομική μας αποστολή στο Αφγανιστάν όπου έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Επίσης η IT προφανώς θα μας απασχολήσει. Ο Καναδάς παίζει σημαντικό ρόλο στην ΑΕΤ και ένα τομέα όπου μπορούμε και πρέπει να ενισχύσουμε τις κοινέ μας προσπάθειες είναι να δούμε το πώς θα συνδεθεί η αντιμετώπιση κρίσεων με τη μακροχρόνια ανάπτυξη, κάτι το οποίο είπα και στην διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την ΑΕΤ την 35η Μαρτίου υπό την κοινή Προεδρία Ένωσης Καναδά, Ισπανίας, Γαλλίας και Βραζιλίας μαζί με τον συνάδελφό μου τον κύριο Πίμπαλξ και την ε, Κρυσταλίνα την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων, χάρηκα για την ανακοίνωση στην ε, Νέα Υόρκη ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ΑΕΤ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν την ενοικοδόμηση της έτης. Επίσης θα δούμε τα της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο μετά την Κομπεχάγη, δηλαδή να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και αυτό σημαίνει πώς θα δούμε και τις πολιτικές ενέργειας θεωρούμε πως η συνεργασία μας με τον Καναδά πρέπει να πάει σε μηχανισμούς χρηματοδότησης και στήριξης της καθαρής ανάπτυξης των τρίτων χωρών. Οι συνέπειε για την Αρκτική είναι άλλο ένα σημαντικό σημείο. Πουθενά αλλού δεν είναι πιο σημαντικές οι συνέπειες αυτές από τη συνεκτική καθώς επηρεάζονται οι άνθρωποι, η βιοπικιλότητα και το τοπίο στη ξηρά και στη θάλασσα. Η προστασία του πληθυσμού της περιοχής είναι βασικός στόχος της ε, πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θα θυμάστε από αυτά τα οποία σας είπα και το Μάρτιο. 40% του εδάφους του Καναδά είναι στον Βορρά, στον Αρκτικό κύκλο, οπότε έχει κοινό συμφέρον μαζί με εμά για την προστασία της Αρκτικής. Τέλος, όσον αφορά τον εξυγχρονισμό της σχέσης μας, έχουμε μια συμφωνία από το 1976, η οποία ισχύει, αλλά είναι πλέον απερχαιωμένη. Θα έχουμε επέκταση της σχέσης μας στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, στη θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών, οπότε χρειάζεται μια άλλη συμφωνία πλαίσιο για να καλύψουμε όλα αυτά τα θέματα, καθώς και μια συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία και για αυτή τη συμφωνία θα συνομιλήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, ε, ζούμε σε έναν κόσμο μεγάλων προκλήσεων και χρειαζόμαστε εταίρους και ο εταίρος είναι ο Καναδάς ένας πιο σημαντικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ κυρία Άστον, δίνω τώρα τον λόγο στην κυρία Γέγλε. Για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Εκπρόσωπε και Αντιπρόεδρε και Βαρόνι κυρία Άστον. Σας ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας είπατε ως ε, αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας με τον Καναδά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι για τη σύνοδο αυτή και για το ότι την συζητάμε. Βεβαίω, όπως ξέρετε, η ψηφοφορία αναβλήθηκε. Δυστυχώς θα ήθελα εγώ όλα αυτά να παρουσιάσω τα σημαντικότερα ζητήματα ε, για εμάς, για το ΕΛΚΑ. Από το 1959 αποτελεί στενό εταίρο της Ένωσης ο Καναδάς. Έχουμε κοινέ αξίες και προσπαθούμε μαζί να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Το 2010 ο Καναδάς ε, είχε την ε, Προεδρία και βεβαίω θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο. Στο πλαίσιο της συνολικής αυτής συμφωνίας είναι σημαντικό να διατηρήσουμε και να εμβαθύνουμε τις καλές μας σχέσεις. Αυτό το οποίο ε, ζητάμε λοιπόν αναφέρεται και στο κοινό μας ψήφισμα ειδικά όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης, ε, την ε, συνεργασία, την αναπτυξιακή, κλίμα, ενέργεια, εμπόριο, οπωσδήποτε και ο γύρος της Δόχας. Βεβαίως ε, τα προβλήματα της καναδικής ευρωπαϊκής ε, πολιτικής καθώς απαιτείται βίζα για πολίτες Τσεχίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας θα πρέπει να αληθούν. Επίσης το άνοιγμα γραφείου βίζα στην Καναδική Πρεσβεία στην ε, Πράγα πρέπει βεβαίως να χαιρετιστούν και η σύσταση ομάδας εργασίας ειδικών και να πω πως είμαι πεπισμένη πως η επόμενη σύνοδος θα επαναβεβαιώσει τις ήδη καλές μας σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την προσοχή σας. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Γέγκλε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τζον Ενσιού. Για δυόμιση λεπτά ακριβώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με προσοχή ακούσαμε αυτά που είπε η κυρία Άστον και συμφωνούμε ότι ο Καναδάς είναι από τους πιο παλαιούς συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η σύνδεση κορυφής ε, ε, που θα λάβει χώρα σε λίγο είναι εξαιρετικά σημαντική για την συνέχιση της συνεργασίας πολλά σημαίνει η σύνοδος αυτή όσον αφορά τη συνεργασία, την ασφάλεια ε, και τις ε, αμοιβαίε συμφωνίες τις οποίες ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε με τον ε, Καναδά όσον αφορά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα για τα οικονομικά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πολύ στενή συνεργασία και στενή συνεργασία επίσης και όσον αφορά την ενέργεια που θα λαμβάνει βεβαίως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε πλευράς, ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά και χρήση φυσικά των τεχνολογιών χαμηλής εκπομπής ε, ρήπων. Συνεργασία όσον αφορά την ε, και άνθρακα. Συνεργασία επίσης ε, όσον αφορά την έρευνα ε, στη, στον ε, Βόρειο Πόλο και γενικότερα συνεργασία όσον αφορά την, τον οικονομικό και πιστοτικό τομέα. Φυσικά θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον Καναδά και όσον αφορά τις πληροφορίες για τους ταξιδιώτες, το PNR. Πιστεύουμε ότι ε, οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα των πολιτών των χωρών μας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ομαλές ε, διμερείς ε, σχέσεις. Αυτή είναι πολύ βασική αρχή και ελπίζομαι ότι και ο Καναδάς από την πλευρά του θα άρει την ανάγκη θεωρήσεων για ορισμένους πολίτες της Ευρώπης. Βεβαίω, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ την ε, σύμφωνη γνώμη που θα πρέπει να δώσει το Κοινοβούλιο ε, για τέτοιου είδου ε, διεθνεί συμφωνίε. και επομένως εξ αρχή θα πρέπει να αναμειχθεί το Κοινοβούλιο με τις διεργασίες αυτής. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ικανοποιητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ενσιού. Βολφ Κλίντσε για 1,5 λεπτό. Κυρίες και κύριοι, οι δύο πλευρές έχουν μια πολύ καλή σχέση, όχι μόνο οικονομική αλλά και συζητήματα εξωτερικών. Σκέφτομαι εδώ πέρα το Ιράν, το Αφγανιστάν, την Αϊτή και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' αυτά έχουμε σοβαρές προκλήσεις μπροστά μας, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε γιατί έχουμε τόσο στενή φιλία. Έχουμε πέντε σημεία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι G20 μίλησαν πολύ και είμαι πεπισμένος πως είναι απαραίτητο στην σύνοδο του Τορόντο, δηλαδή υπό καναδική ηγεσία, να δούμε πώς θα έχουμε αποτελέσματα και όχι μόνο υποσχέσεις. Δεύτερον, αναφέρθηκε κλιματική πολιτική. Έχουμε παρόμοιους στόχους. Εμείς μπορούμε να διδαχτούμε από τον Κάναδα το τι γίνεται με τον δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Τρίτον, χρειάζεται μια νέα εμπορική συμφωνία και εδώ πέρα νομίζω πως οι στόχοι μας είναι πάρα πολύ κοντά. Δύο πράγματα θα ήθελα να παρατηρήσω, που υπάρχει καλή πρόθεση αλλά ακόμα δεν έχουμε πλησιάσει. Πρώτα απ' όλα για την βίζα, το αναφέρατε κύριε Πατή εκπρόσωπε, ελπίζω πράγματι να τα καταφέρουμε να μεταχειριστούμε με τον ίδιο τρόπο εθνικές μειονότητες από κράτη-μέλη της Ένωσης και δεύτερον συμφωνία για τα δεδομένα αεροπορικών επιβατών. Ε, ισχύει de facto αλλά χρειαζόμαστε μια νέα νομική βάση για να εξακολουθεί να ισχύει και να διασφαλίζει πως αυτά τα οποία έχουμε εμείς ως δικαιώματα να ισχύουν και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι δυνατόν πλέον όλες αυτές οι πληροφορίες όνομα, γενέθλια, πιστοτικές κάρτες να πηγαίνουν και να τα κάνουν καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να δημιουργηθεί μια νομική βάση που θα ανταποκρίνεται και σε αυτό το οποίο θα είναι και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κλίντς. Ο κύριος Μπουτικόφερ τώρα. Για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, ο Καναδάς για εμάς είναι ένας καλός φίλος, σημαντικός εταίρος, σημαντικός διεθνής εταίρος και είναι μια όρημη δημοκρατία από την οποία μπορούμε να μάθουμε πολλά. Αλλά ειδικά όταν ξέρουμε πως ε, έχει αποφασιστεί εδώ πέρα ψήφισμα περί Καναδά να το παίρνουμε πιο σοβαρά και να ασχολούμαστε σοβαρότερα με τις ευρωκαναδικές σχέσεις από ό,τι είναι η προσπάθεια στο υποβληθέν ψήφισμα. Δεν, εγώ δεν νιώθω άνετα. Από τις, μιλάμε για κοινέ προκλήσεις, αλλά δεν αναφέρεται καν η Αρκτική. Δεν αναφέρεται η προστασία της Αρκτικής, παρά μόνο σε μια δευτερεύουσα πρόταση. Σουηδία, Ισλανδία, Φιλανδία δεν ε, προσεκλήθησαν από τον Καναδά στην σχετική συνάντηση. Επίσης δεν αναφέρεται το πετρέλαιο που θα αντληθεί από τα αμμώδη εδάφη. Επίσης τι γίνεται με τον ε, ερυθρό τόνο. Δεν θα έλεγα πως προκαλεί ο Καναδάς, αλλά αν να μιλήσουμε ειλικρινά μεταξύ φίλων δεν είναι σωστό να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Λένε πως ο Καναδάς δεν έπαιξε σοβαρό ρόλο, δεν έπαιξε θετικό ρόλο στην Κοπενχάγη και πως το πρόβλημα της βίζας με την Τσεχία και τους Ρωμά με την Τσεχία πρέπει να το τονίσουμε. Οπότε, να συνεργαστούμε φιλικά, αλλά να μην ξεχνάμε τις δυσκολίες, δεν εξυπηρετούμε κανέναν. Γι' αυτό η δική μου ομάδα θα ζητήσει όταν θα ψηφίσουμε να δούμε τα προβλήματα του πετρελαίου από την άμμο από τα αμμόδια έδαφα και από τα αμμόδια έδαφα με και τα άλλα προβλήματα που ανέφερα. Now the floor to Philip ε, Bradburn. Ευχαριστώ το λόγο και ο κύριος Μπράντμπουρν. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής για τη σχέση με τον Καναδά, καλωσορίζω αυτό το ψήφισμα. Είναι το πρώτο για το, μετά τον διάσκεψη. Ο Καναδάς είναι ο αρχαιότερος ε, εταίρος μας ε, και έχει αποτελέσει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, είπε και η κυρία Άστον, οι διαπραγματεύσει προοδεύουν με τον Καναδά για μια συνεκτική συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει αυτές, αυτή τη συμφωνία και ελπίζω η Κομισιόν να μας κρατήσει ενήμερους για όλες τις εξελίξεις και σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων. Το ψήφισμα που έχουμε ενώπιόν μας ε, το υποστηρίζουμε διότι είναι σύντομο και αφορά τα σημαντικά ζητήματα των διαπραγματεύσεων με την κανονική κυβέρνηση. Αποτελεί μια επαρχή για τι μελλοντικέ διαπραγματεύσει και δείχνει ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να έχει πιο στενές σχέσει με έναν ε, παλαιό εταίρο. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε όχι μόνο τις σχέσεις μας ως Κοινοβούλιο, αλλά και την συνεργασία μας με τρίτες χώρες. Ευχαριστώ κύριε Μπραντμπορν. Το λόγο έχει ο κύριος Higgins για δυόμιση λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, δεν είχαμε καμία αξιολόγηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αντικτύπων αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Η Καναδική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων με 600.000 μέλη που δουλεύουν σε δέκος μεταφορές, σε νοσοκομεία, ανησυχεί για τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας. Η Εθνική Ένωση ε, υπαλλήλων στον Καναδά με 340.000 μέλη, Ένωση Ιδιωτικού Τομέα με 60.000 μέλη στον τομέα της υγείας ανησυχούν. Γιατί, Γιατί φοβούνται πως ε, θα εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των εργαζομένων ή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και η ευρωπαϊκές ε, και οι καναδικές πολυεθνικές θέλουν να μπουν στην παροχή κοινοφελών υπηρεσιών και θεωρούν πως η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά θα σημάνει ιδιωτικοποίηση του νερού, των μεταφορών και του ηλεκτρισμού. Καταστροφικό αυτό για τον μισθό των Καναδών εργαζομένων καθώς θα μειωθεί πάρα πολύ όπως είδαμε και στην Ευρώπη. Η δε ίδια η Κομισιόν υποστηρίζει τα δικαιώματα των εταιριών για να εκμεταλλεύονται τους εργάτες. Όπως αποδεικνύεται από το ότι έσυρε το Λουξεμβούργο στο δικαστήριο γιατί προσπάθησε να δώσει τα ίδια δικαιώματα στους μετανάστες με τους Λουξεμβούργιους. Και τι θα κάνουν τώρα, θα ιδιωτικοποιήσουμε το νερό στον Καναδά. Μην ξεχνάτε τι έκαναν ευρωπαϊκέ πολυεθνικέ στη Βολιβία με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ευτυχώ, οι φυσιολογικοί άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι στον Καναδά είναι διατεθειμένοι να παλέψουν για το νερό του. Και οι ενό του δημοσίου τομέα στον Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν και θα πρέπει να ξεκινήσει μια εκστρατεία για να προστατευτεί η δημόσια διοικησία των δημοσίων και κοινοφιλών υπηρεσιών και όχι μόνο να υπάρχει στο στόχος ε, η μεγιστοποίηση των κερδών. Και δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για συνόδους κορυφής, πρέπει και απλοί άνθρωποι να συναντηθούν να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Ρόσμπαχ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρε, η Ευρώπη και ο Καναδάς συνεργάστηκαν άψογα τον τελευταία, χρόνια και γι' αυτό προσβλέπουμε σε μια περαιτέρω συνεργασία. Τώρα, αν διαπραγματεύσεις ε, καθυστερούν, τότε διαδικασία την οποία ακολουθούμε ίσως να είναι πάρα πολύ χρονοβόρο. Ίσως ε, με άλλο τρόπο θα μπορούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει παραδείγματος χάρη το θέμα της απαγόρευσης ε, κυνηγιού της ε, φώκιας που αντιβαίνει όλων των συμφωνιών για την προστασία των ζώων αλλά και το ζήτημα των μεταφορών, η μετάβαση από τον βόρεια στα βορειοανατολικά ανατολικα βορειοδυτικά που είναι ένας τρόπος ε, για την εξοικονόμηση ενέργειας, ε, καυσίμων και την βελτιστοποίηση των ε, μεταφορών. Καθώς επίσης και η απαγόρευση για την διέλευση δεξαμενοπλοίων στην ανοιχτή θάλασσα. Το λόγο έχει ο κύριος Μόλτσαρ. Κύριε Πρόεδρε, σαν να μην έφτανε πως στη μέση των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας προέκυψαν πληροφορίες που έλεγαν πως ο Καναδός στο πλαίσιο της ε, ΣΕΤΑ και της ΑΚΤΑ θα προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό και αμερικανικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας φαίνεται πως πηγαίνουμε και προς την κατεύθυνση έντονων ιδιωτικοποιήσεων. Βεβαίως Εντάξει, να δίνονται μεγάλα συμβόλαια και να υπάρχουν οι ανάλογοι κανόνες για να μην υπάρχει διαφθορά κτλ. Αλλά όταν παραπονιούνται ήδη εδώ πέρα οι δικοί μας οι δήμοι για το ότι είναι αναγκασμένοι να ευνοούν τεράστιες επιχειρήσεις, ε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να το κάνουν αυτό και άλλες χώρες και όταν αποφασίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις τις πολιτικές για το περιβάλλον και μπορούν μετά να ζητήσουν και αποζημίωση με βάση αυτές τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου φαίνεται πως δεν έχει δαχθεί τίποτα από την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν είναι πραγματικά να ωφελήσει τους πολίτες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελέσει προπύργιο κατά της παγκοσμιοποίησης. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Κριστιαν Πρέντα για ένα λεπτό και δεκατρία. δε, και δεύτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρωτίστως ε, να τονίσω πως ε, η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά είναι ε, μια πολύ σημαντική συνάντηση προκειμένου να εμβαθύνουμε περαιτέρω τις σχέσεις που έχουμε με αυτήν την μεγάλη δημοκρατία. Οι σχέσεις μας είναι πολύ σημαντικές τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που ο Καναδάς έχει τις ίδιες αξίες με εμάς και συνεργάζεται εδώ και πολύ καιρό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπενθυμίσω επίσης ε, πως ε, μετά από τη διακήρυξη τη προηγουμενη διάσκεψη διαθέτει της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά που διεξήχθη τον Μπράγα τον Μάιο του 2009 θέσαμε στου στόχους ε, ότι δηλαδή οι εταίροι θα πρέπει να μαθαίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία, ελεύθερη διακίνηση προσώπων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια περιοχή ε, κυκλοφορίας ε, και διακίνησης δίχως ε, προξενικές θεωρήσεις. Ένα χρόνο αργότερα πρέπει να πούμε ότι αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθηκε. Ρουμάνοι, Βούλγαροι χρειάζονται προξενική θεώρηση για να μεταβούν στον Καναδά αλλά επαν άρχισε να επανισχύει η θεώρηση και για τους ε, Τσέχους πολίτες. Εδώ υπάρχει ζήτημα αμοιβαιότητας, διότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν καταργήσει την βίζα για τους Καναδούς πολίτες και υπάρχει και ένα ζήτημα συνέπειας, διότι αφενός ο Καναδάς κατήργησε τις ε, θεωρήσεις για την, από την Κροατία μάλλον που είναι μια χώρα υποψήφια αλλά συνεχίζει να διατηρεί τις θεωρήσεις για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάσκεψη κορυφής θα πρέπει να ε, ρυθμίσει αυτό το ζήτημα προκειμένου να καταργηθούν οι θεωρήσεις για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται να θέσουμε αυτό το ζήτημα πολύ ψηλά στη μεσαιτιάταξη. Δεν είμαστε διόλου... Ε, ικανοποιημένοι από τις ε, διακηρύξεις ε, αρχών. Αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ε, πολίτες της χώρας μου, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Το λόγο έχει ο κύριος Λάιχφριντ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι γιατί έχω πάντα την αίσθηση πως πρέπει να υποπτεύομαι την Κομισιόν πως δεν θέλει να φέρει πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ίδιο ισχύει και για την Συμφορία Ελευθερίου Εμπορίου με τον Καναδά. Θα συμφωνήσω εδώ με τους συναδέλφους που λένε πως υπάρχουν κάποιες υποψίες, ειδικά σχέση με αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Χίγκινς και του δίνω απολύτως δίκιο. Οι συμφωνίες εμπορίου, κατά την άποψή μου, είναι θετικές όταν προωθούν αμοιβαία την ευημερία και όχι όταν ε, αποκλειστικά εξυπηρετούν τα συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών. Και όταν λαμβάνουμε πληροφορίες πως σε μια τέτοια συμφωνία η υγεία, η εκπαίδευση, η δημόσια τάξη ξαφνικά είναι αντικείμενο εμπορίου και πρέπει να απορριθμιστούν και να ιδιωτικοποιηθούν, τότε έχω την υποψία πως τι έχουμε εδώ πέρα, κέρδος των ολίγων και ζημία των πολλών. Αυτά τα πράγματα έρχονται ως συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, όταν διαπραγματευόμαστε με έναν εταίρο όπως ο Καναδάς, πρέπει να αναφέρουμε και ορισμένα πράγματα που δεν είναι τόσο ευχάριστα και που πρέπει να υποθούν. Π.χ. η σφαγή των μικρών φωκιών. Όχι μόνο για να εκνευρίσουμε κάποιον, για να ξεκαθαρίσουμε την ευρωπαϊκή στάση, για να βρούμε μία λύση για αυτό το ε, φρικτό ε, εμπόριο εις βάρος μικρών ε, ζώων. Ευχαριστώ. πάρα πολύ κύριε Λάιχτφριντ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο συνάδελφος Σεμπαστιάν Μπουντού δεν, μπορούσε, δεν μπόρεσε να φτάσει στο Στρασβούργο, γι' αυτό λοιπόν μιλάω εξ του. Αυτή τη στιγμή 3,9 εκατομμύρια πολιτών της Ευρώπης δεν μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς θεώρηση, χωρίς βίζα δηλαδή, στον Καναδά ο Καναδάς και οι Ηνωμένε Πολιτείε κρατούν, διατηρούν αυτήν την θεώρηση δημιουργώντας ε, πολίτες Ευρωπαίους ε, δύο ταχυτήτων και δημιουργώντας βεβαίως προβλήματα. Ο πρόεδρος ε, Μπαρόσο στην προηγούμενη διάσκεψη κορυφής επέμενε στην επίλυση του προβλήματος αυτού και πρέπει να διατηρήσουμε την ίδια, να επιμείνουμε στην ίδια στάση. Από το 2004 τα αιτήματα ε, των ε, Ρωμάνων πολιτών μειώθηκαν από 16% σε 5% ε, και οι περισσότεροι έχουν ενταχθεί σε επίσημα μεταναστευτικά προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω γιατί ο Καναδάς το 2009 ε, σταμάτησε να απαιτεί ε, θεώρηση για, για πολίτες ε, υπό ένταξη χώρας, υποψήφιας χώρας, ενώ, δεν, ενώ εξακολουθεί να ζητά θεώρηση από τους Ρουμάνους πολίτες. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν ε, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο επανειλημμένα έχει θίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, είναι μια απόφαση ήδη του 2009 που θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να διατηρηθεί και να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αλληλεγγύη σε περίπτωση που το πρόβλημα αυτό δεν λυθεί μέχρι του χρόνου. Αυτό η Λεδιάστον θα πρέπει οπωσδήποτε να το λάβει υπόψη της. Ευχαριστούμε πολύ. Μουτσουμέσκλη, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινέσκου. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Αρσένη, στον κύριο Κρήτονα Αρσένη για 1,5 λεπτό. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Καναδά είναι ένα από του πιο παλιού και στενού συμμάχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από το 1959. Ωστόσο, η συνεργασία μα πρέπει πάντοτε να στηρίζεται σε κοινέ αξίε και αμοιβαίο σεβασμό ο καναδά είναι μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων ρηπαντών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίω και είναι η μοναδική χώρα που ενώ υπέγραψε και κύρωσε το πρωτόκολλο του κιότο στη συνέχεια ανακοίνωσε δημοσίω ότι δεν έχει σκοπό να τιμήσει τι νομικέ δεσμεύσει τη. αντί να μειωθούν οι εκπομπέ του κατά 6 σε σχέση με το 1990 οι εκπομπέ του καναδά αυξήθηκαν κατά. 26 η παραγωγή πετρελοφόρου άμμου είναι η βασικότερη αιτία. Η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή πετρελοφόρου άμμου είναι τρει έω πέντε φορέ μεγαλύτερη από εκείνη τη συμβατική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου η παραγωγή περιτρελοφόρου άμμου απαιτεί επίση δύο έω πέντε βαρέλια νερό για κάθε βαρέλι πίσας που εξάγεται και στη συνέχεια δημιουργεί μια σειρά αποβλήτων που απειλούν τόσο την βιοποικιλότητα όσο και τη ζωή των ηθαγενών. η παραγωγή επίση αυτή καταστρέφει το δάσο Μπορέαλ, μία από τι μεγαλύτερε δεξαμενέ άνθρακα στο πλανήτη. μέχρι το 2020 η πετρελαιοφόρος άμμος μάλλον θα παράγει περισσότερε εκπομπέ από ότι η αυστρία και η ιρλανδία ο καναδά ξοδεύει μόνο εβδομήντα δολάρια ανά άτομο για πράσινε ενισχύσει την ίδια στιγμή που η κορέα ξοδεύει χίλια η αυστραλία 420 και η ηπα. ΕΕ 365. η διασφάλιση τη προστασία του δάσου boreal είναι πάρα πολύ σημαντική ε, και είναι σημαντικό να ζητήσουμε από τον καναδά να συμμορφωθεί με τι διεθνεί συμφωνίε που έχουμε από κοινού υπογράψει αλλά μόνο μονομερό σεβόμαστε εμείς και αυτό θα πρέπει να είναι βάση για όποια περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ατσένη. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μύροσλαβ Μικολάζικ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Αντιπρόεδρε. Από το 1959 ο Καναδάς είναι ο πιο κοντινός και ο πιο σταθερός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που η σημερινή δεξιά κυβέρνηση καταφέρνει το οικονομικό της έργο και την οικονομική ανόρθωση του Καναδά διορθώνοντας λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης. Η οικονομική κατάσταση βελτιώνει και την κατάσταση του δολαρίου και το βιωτικό επίπεδο των Καναδών δημιουργεί επομένως και καλές προϋποθέσεις για την πολιτική και κυρίως οικονομική συνεργασία με άλλες χώρες. Είναι πεπισμένος ότι η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά στις Βρυξέλλες θα δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω προώθησης της συνεργασίας και κυρίως της οικονομικής εταιρικής σχέσης. Ο Καναδάς είναι ο ενδέκατος στη σειρά σημαντικότερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύει 1,7% ε, ε, του εξωτερικού εμπορίου και ο Καναδάς είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος επενδυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 49,9 δις ευρώ σε αγαθά ανταλλάχθηκαν το 2008 και αντιστοίχως 20 δις αντιπροσωπεύουν οι υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι σχέσεις με τον Καναδά είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις, εποφελία και των δύο πλευρών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζωάν Βρεζινά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπο, η πολιτική εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και υπάρχει αυτό το θέμα των θεωρήσεων για παραδείγματος χάρη ε, των ε, Τσέχων πολιτών για την μετάβασή του στον Καναδά. Εμείς ως Τσέχοι θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Πραγματικά παραβιάζονται τα δικαιώματα των ε, πολιτών και παράλληλα το κύρος των ευρωπαϊκών θεσμών το οποίο απειλείται η θέση της καναδικής κυβέρνησης Νομίζω ότι προσβάλλει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρεάζει τη συνοχή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να ε, υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη και τα συμφέροντά τους. Η τελευταία ευκαιρία που θα έχουμε θα είναι αυτή η συνάντηση, η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Θα πρέπει να τεθεί αυτό πολύ ψηλά στην μέσα διάταξη της εν λόγω διασκέψεως. Το ζήτημα θα πρέπει να επιληθεί από το 2009 όταν ε, εγκρίθηκε πως ε, θα πρέπει να ε, καταργηθούν οι θεωρήσεις ξέρουμε ότι ένα τμήμα της συμφωνίας εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατόν να δεχτεί κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να δράσει και θα πρέπει να λάβει θέση και να ζητήσει από τον Καναδά να σεβαστεί τα συμπεφωνημένα. Θεωρώ πως ε, η κατάσταση θα πρέπει να τελειώσει. Οι Τσέχοι πολίτες αυτό προσδοκούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν ε, περιμένουν λόγια, περιμένουν συγκεκριμένες δράσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. ο οποίος ε, θα παρευρεθεί στην διάσκεψη, χρειάζεται να δράσει. Πρέπει λοιπόν ε, να ενεργήσουμε με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό. Ε, εάν δεν πετύχουμε αυτό το οποίο προσδοκούν οι πολίτες μας, τότε θα αφηγεί το κύρος μας. Εν ώψη στο της λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε στην στο αίτημα για τον σεβασμό αυτής της συμφωνίας. Το λόγο του κ. Κάρας. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ω μέλο της αντιπροσωπείας με τον Καναδά πρέπει να τονίσω πως έχουμε κοινέ αξίες με τον Καναδά. Οι κοινέ μας αξίες είναι θεμελιώδης για την διαμόρφωση της κοινωνίας μας. Αυτή η κοινή βάση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε τις παγκόσμιες συνθήκες. Οι στενές ιστορικές και πολιτισμικές σχέσεις, όπως και ο σεβασμός για την πολυμέρεια και την χάρτα του ΟΗΕ αποτελούν τη βάση της εταιρικής μας σχέσης. Πρέπει να βελτιώσουμε τα διάφορα επίπεδα των σχέσεών μας και οπωσδήποτε και το πολιτικό. Με την σημερινή συμφωνία για πρώτη φορά έχουμε μια συμφωνία με βάση τη νέα μας συνθήκη. Πρέπει να το ξέρει αυτό η Κομισιόν. Διαφάνεια, συνεργασία, εμπλοκή του Κοινοβουλίου είναι προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτή η συμφωνία. Και έχουμε δύο σημαντικά θέμα. Η μονομερής επιβολή βίζας κατά των Τσέχων ε, συμπολιτών μας, η οποία είναι ανεπίτρεπτη. Η κριτική δε του Καναδά για την ε, συμφωνία και για τις προϋποθέσεις που τίθενται σε ορισμένα προϊόντα δείχνει πως πρέπει να αλλάξει ο Καναδάς και όχι εμείς και πράγματι ο Καναδάς είναι, βεβαίω μέλο, βεβαίως μέλος και στην ναύτα και αυτό νομίζω αποτελεί και ένα μήνυμα κατά του προστατευτισμού και είναι ωραίο μήνυμα το ότι την ημέρα που θα έρθει ο Τζο Μπάιντεν στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε και την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά γιατί έχουμε νομίζω συνεργασία η οποία είναι σημαντική και με τις δύο χώρες της ε, Βορείου Αμερικής εάν θέλουμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάρας. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Ρόιτοβα. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, θα ήθελα να πω ότι αυτή η μονομερής απέτηση βίζας ε, για τους ε, πολίτες τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα αποτελέσει και την αχίλιο πτέρνα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με τον Καναδά. Ο Καναδάς θα πρέπει να προσαρμόσει και την νομοθεσία του περί ασύλου. Η Λεβιάστον Μάλλον, ε, ε, σας ερωτώ, ε, Λέδη Άστον, σημειώσατε στον Καναδά ότι αυτό το 2030 δεν είναι ικανοποιητικό έτσι ώστε ο Καναδάς να αποτελέσει χώρα ε, για τους ετούντες άσυλο. Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει οπωσδήποτε επισταμένος να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα των ταξιδιωτικών θεωρήσεων. Γιατί διαφορετικά φαντάζομαι ότι γνωρίζετε τον κίνδυνο ε, μη υπογραφής της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί βεβαίως δεν πρόκειται εμείς να δεχτούμε μονομερή δράση εναντίον τριών χωρών. Χαίρομαι που στο ψήφισμά μας ε, υπάρχει σαφής αναφορά ε, στις ε, θεωρήσεις και στην προσαρμογή της πολιτικής του Καναδά όσον αφορά το άσυλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ροϊτόβα. Θα ξεκινήσουμε... Λέει ο, κύριος, λέει ο Πρόεδρος στη διαδικασία Catch the Eye, ο κύριο Σιλβέστρης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπο, η συζήτηση ε, στην ε, Ολομέλεια βεβαίως σας δυναμώνουν εν ώψη της διάσκεψη κορυφή του Μαΐου. Αναμφίβολα οι αρχές που εκφράστηκαν εδώ ε, όλες συγκλίνουν στην σημασία που αποδίδουμε στη συνεργασία μα με τον Καναδά. Πρόκειται για μια μεγάλη δημοκρατική χώρα ναι, και είναι στρατηγικό μα συμφέρον να έχουμε σχέσεις με τη χώρα αυτή. Υπάρχουν όμως και μεμονωμένες ε, προτάσεις, μεμονωμένα προβλήματα τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να αντιμετωπίσετε και ενδεχομένως να λύσετε στο μέτρο του δυνατού στη διάρκεια της διασκέψης κορυφής. Γιατί αποτελούν αιχμή δόρατος πολλών ε, θεμάτων. Αυτή η αρχή της αμοιβαιότητας όσον αφορά την κυκλοφορία των Καναδών και Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ δεν είμαι ούτε Ρουμάνος, ούτε Βούλγαρος, ούτε ε, τσέχο. Αλλά εγώ είμαι Ευρωπαίος πολίτης και επομένως πραγματικά αισθάνομαι εξαπατημένο. Ε, πραγματικά αισθάνομαι ότι ε, Κοιτάξτε, εγώ μιλάω γρήγορα, ε, γιατί με καταλαβαίνετε κύριε Πρόεδρε. Α, υπάρχει και η διερμηνία, ναι, έχετε δίκιο. Να μιλάω λίγο πιο αργά λοιπόν. Ωραία, <laughs> λοιπόν, υπάρχουν ε, ε πολίτε ε, οι οποίοι μπορούν ε, χωρί κανένα πρόβλημα να κυκλοφορήσουν στον Καναδά, ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Αντιθέτω, όλοι οι Καναδοί πολίτε μπορούν ε, ανεξαρτήτω χώρα να κυκλοφορήσουν στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης βλέπουμε από μελέτες, βλέπουμε και στην τηλεόραση κάποιες ε, εκπομπές, ε, κάποιους τρόπους κυνηγιού ε, που μας δημιουργούν συναισθηματικά προβλήματα. Μας προβληματίζουν λοιπόν οι εικόνες που βλέπουμε, αλλά από τη συγκίνηση και από το συνέστημα θα πρέπει και από τα λόγια, θα πρέπει να περάσουμε τώρα στις πράξεις, να κάνουμε κάτι και να ζητήσουμε πάυση αυτού του είδους κυνηγιού. Ε, θα θέλαμε επίσης, ε, κυρία Επίτροπε, να αναφερθείτε μετά στο Κοινοβούλιο, ενώ μετά από τη διάσκεψη κορυφής του Μαΐου. Ευχαριστώ κύριε Σιλβέστρη. Το λόγο έχει η κυρία Όλγα Σεμαλόβα. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από την Σύνοδο με τον Καναδά θα ήθελα να υπενθυμίσω μια από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αρχή της αλληλεγγύης είναι μια από τις αξίες που πρέπει να γίνεται συνεχώς σεβαστή εάν είναι να είναι αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν μία μόνο χώρα έχει δυσκολία πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Όπως είπαμε τον Ιούλιο του 2009 ο Καναδάς επέβαλε υποχρέωση βίζας στους Τσέχους πολίτες κατόπιν αιτήματος της ε, Τσεχικής Δημοκρατίας το Συμβούλιο Εσωτερικών έθεσε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του Φεβρουαρίου παρά το έργο διαφόρων ομάδων ειδικών και την στήριξη κρατών μελών δεν έχει υπάρξει αυτή πρόοδος το τον αναμένουμε τώρα πιθανές αλλαγές ε, στον κανονισμό το 2013 δεν προσφέρει τίποτα στους ε, Τσέχους ε, πολίτες. Συχνά μιλάμε για την κρίση εμπιστοσύνης έναντι των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και νομίζω πως κάτι καλύτερο πρέπει να κάνετε και εσείς κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ τον λόγο ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω, είπατε εκπρόσωπος, να συγχαρεί τους Καναδούς για τη διπλωματία τους, γιατί έχουν αρκετά να μας διδάξουν. Στην τελευταία διάσκεψη για το εμπόριο απειλουμένων ειδών συμμάχησαν με τους Ιάπωνες για να μας νικήσουν πλήρως όσον αφορά τον ερυθρό τόνο. Κάτι το οποίο βεβαίως μας θύμισε την Κοπενχάγη όπου ήταν ασαφής η θέση της Ένωσης, συζητούσαμε μεταξύ μας αντί για να συζητάμε με τους άλλους καθημερινά και καταλήξαμε να μας ισοπεδώσουν. Η Απονία και ο Καναδάς επί ε, ασκούσαν επιρροή για να βρουν τις ψήφους που ήθελαν, για να κάνουν αυτό που ήθελαν. Και εμείς πάλι ασυντόνιστοι ήμασταν και ανοργάνωτοι και αδύναμοι ο ε, Επίτροπος Περιβάλλοντος είπε πως δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Αλλά διασκέψεις τέτοιες γίνονται συνεχώς ανά τον κόσμο και πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως την διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε μια στρατηγική για το μέλλον, να χρησιμοποιήσουμε σωστά τους πόρους μας και να μην ε, έχουμε λιγότερο ειδικό βάρος από αυτό που μας αναλογεί. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Σόμπερ θα ήθελα να φερθώ σε ένα δύσκολο πρόβλημα για τα δικαιώματα κάποιων συγκεκριμένων αγαθών. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με κάποιους καθηγητές όσον αφορά το copyright και τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. θα υπάρξει πλήρης αναθεώρηση του σχετικού ε, καναδικού δικαίου και βεβαίως από την άλλη απαιτούνται ειδικά όσον αφορά την προστασία από αντιγραφή ε, των ε, ταινιών και οπτικοακουστικών προϊόντων πολύ αυστηρές διατάξεις. Αυτό έχει βεβαίως μεγάλη σημασία και να υπάρξει και συμπερίληψη του διαδικτύου καθώς αυτό ακριβώς καθιστά αδύνατη την προστασία τέτοιων αγαθών εάν δεν υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες. Ε, να υπενθυμίσω εδώ πέρα την απαγόρευση βιντεοκαμερών που, στους κινηματογράφους που πρέπει να εφαρμοστεί και στον Καναδά. Εντάξει, προστασία αλλά όχι και πλήρη επιτήρηση του ίντερνετ. Βλέπουμε επίσης πως ο Καναδάς έχει και διαφορετική νομική παράδοση και ε, σύστημα, οπότε ελπίζω να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο. Σας ευχαριστώ κύριε Ομπερμάερ. Λόγο τώρα έχει ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω πως το σημαντικότερο εδώ πέρα είναι να δώσουμε βάρος μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί βρισκόμαστε σε μια οικονομική κρίση και τις 100 των φορολογικών εσόδων προέρχονται από αυτές. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δημόσιες προμήθειες να επικεντρωθούν στο να αποκτήσουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυνατότητα να χτυπήσουν τέτοια συμβόλαια. Και βεβαίως χρειαζόμαστε και τις τεχνικές προδιαγραφές, αυτό το οποίο λέμε trade facilitation, σε αυτή την συμφωνία. Το ερώτημά μου είναι Υπάρχει εδώ πέρα με τον ΠΟΕ μια κοινή συμφωνία έτσι ώστε οι βάσεις ε, των διαπραγματεύσεων να ε, ληφθούν υπόψη στην συμφωνία αυτή ελευθεροπορίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Ευχαριστώ πολύ η Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, το ζήτημα αυτό είναι ζωτική σημασία προκειμένου να μπορέσει ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθουν ακόμα πιο κοντά. Η συμφωνία που είχε συναυθεί για τις αεροπορικέ μεταφορές ε, τον Δεκέμβριο 2009 και η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά αναφορικά με την ασφάλεια των ε, πτήσεων που υπογράφει και αυτή το 2009 είναι δύο σημαντικά στοιχεία των ε, σχέσεών μας. Η πρώτη είναι προσωρινού χαρακτήρα μέχρι την ε, οριστική επικύρωσή της. Ε, το Καναδάς δεν έχει λάβει καμία επιβεβαίωση πάνω σε αυτό. Το, το δεύτερο, η δεύτερη όμως δεν είναι προσωρινή. Το Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλει μια σαφή και συγκεκριμένη πρόταση τώρα σε ό,τι φορά την συνεργασία μας θα, θα σας ζητήσω κυρία Αντιπρόεδρε πότε οι δύο αυτές συμφωνίες πρόκειται να ισχύσουν ουσιαστικά αναφορικά με τις αεροπορικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Φιώνα Αλ. E Ο Καναδάς είναι στενός φίλος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι κριτικός φίλος όταν ε, είναι ε, απαραίτητο. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Κοπενχάγη ε, ε, ξέφυγε ε, η, ο Καναδάς και όπως είπε και ο κ. Αρσένης το ζήτημα της πετρελοφόρου άμμου είναι πάρα πολύ σημαντικό και οπωσδήποτε εξαιρετικά ρηπαντικό. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια ε, πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να μειωθεί η ισχύ της ε, οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον Καναδά ε, να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Χαουλ. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Άστον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και ε, ωφέλιμη ε, συζήτηση γιατί εκαλύφθησαν μια ε, ευρεία σειρά θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Πρόκειται για θέματα τα οποία βεβαίω έχει υπόψη τη και η Επιτροπή και το Συμβούλιο και όσοι θα ηγηθούν τη διασκέψεω κορυφή. Παρ' όλα αυτά, είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων προ όλου όσου εξέφρασαν τα συγκεκριμένα ε, σχόλια ε, και τα οποία θα μας ε, βοηθήσουν. Βεβαίως υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να σας απαντήσω εδώ όσον αφορά ας πούμε τις για τους επιβάτες κλπ. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι όλοι οι βουλευτές ε, κρίνουν σημαντική την συνεργασία με τον Καναδά ε, και επίσης κρίνουν σημαντικό το στοιχείο ε, του, της συνεργασίας και της, των αρχών που χαρακτηρίζουν και τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι έχουμε δίκιο που προσβλέπουμε σε μια φιλόδοξη εμπορική συμφωνία και νομίζω ότι και από τη μικρή και νομίζω ότι και από την αρχή ε, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, της, ε, των εμπορικών συμφωνιών Καναδά Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν πρόκειται για εύκολες συζητήσεις. Τα, ε, βεβαίως το θέμα της εξόρυξης ε, ασφαλτικής άμμου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι κάτι εξαιρετικά ε, σημαντικό και προχωράνε όμως οι συζητήσεις αυτές. Βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, ε, θα πρέπει να μελετήσουμε από κοντά όλα τα ε, θέματα και μάλιστα σε λεπτομέρεια και βεβαίως το Κοινοβούλιο θα παίξει τον ρόλο του έτσι ώστε να συμφωνήσει με την ε, πρόταση συμφωνίας που θα του υποβληθεί. Θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα. Πρώτον, μια καλή εμπορική συμφωνία είναι επωφελής προς όλους τους πολίτες. Είναι καλό για τους καταναλωτές, δίνει ευκαιρίες στους εργαζόμενους και βεβαίως όλες οι εμπορικές συμφωνίες μας δίνουν πραγματικές ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις στατιστικές που πάντοτε με εξέπληταν είναι αυτό το 8% των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας που έχουν ανταλλαγές με χώρες εκτός των συνόρων και 3% με χώρες εκτός, έχουν επαφές δηλαδή με χώρες εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν υπάρχει μεγάλο πεδίο ευκαιριών συνεργασιών και από τις δύο πλευρές που θα είναι επωφελή συνεργασία συνεργασία προς όλους. Βεβαίως ε, αρκετά μέλη ε, αναφέρθηκαν ε, στο θέμα των ερευνών στην Αρκτική. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και γιατί σχετίζεται και με άλλα σημαντικά θέματα, όπως πούμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Είναι γεγονό ότι ο Καναδάς στη διάσκεψη τη Κοπεχάγης, κατά την άποψή μα τουλάχιστον, ήταν μέρο των χωρών αυτών που δεν βοήθησαν ιδιαίτερα στο να προωθηθεί ο διάλογο. και ελπίζουμε θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε. Επίσης, την 3η Μαρτίου είναι σαφές ότι η Καναδέζικη κυβέρνηση δήλωσε ότι ο Καναδάς θα ακολουθήσει τις αποφάσεις της ε, Κοπενχάγης. Βεβαίως ε, θα πρέπει να πιέσουμε ε, τον Καναδά έτσι ώστε να, να πιέσουμε λέω τον Καναδά έτσι ώστε τουλάχιστον να συμφωνήσει με, την, τον μετριασμό των εκπομπών βάσει της συμφωνίας 20 green 2020 ε, και να ενισχύσει την χρήση πράσινης ε, τεχνολογίας και όλα αυτά τα μέτρα ε, μετριασμού των εκπομπών των οποίων συμφωνούμε και τα οποία αναφέρονται στην στρατηγική 2020. Το άλλο θέμα, το θέμα των ταξιδιωτικών θεωρήσεων βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Τρεις είναι οι χώρες μέλη οι οποίες επηρεάζονται από την απόφαση του Καναδά όσον αφορά τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις. Βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει ε, να συζητηθούν, τα οποία αφορούν το μέλλον ε, και που είναι νομοθετικού περιεχομένου. Νομίζω ότι η δεύτερη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα εργαστεί στην Τσεχία έτσι ώστε να δει από κοντά το τσεχικό ζήτημα και βεβαίως θα εργαστεί η ομάδα αυτή υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Χαίρομαι που θίγονται τα ζητήματα αυτά και τα οποία βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα και υπενθυμίζω ότι δεν πρόκειται για διμερεί ζητήματα, είναι ζητήματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά και σαν τέτοια θα αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Άστον, ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο στη συζήτηση αυτή η οποία μόλις ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία επί της συζητήσεως αυτής θα λάβει χώρα στην επόμενη σύνοδο Ολομελίας. Ε, θα διακόψουμε για την ώρα, θα ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας στις 19 ακριβώς με την ώρα ερωτήσεων προς την Επιτροπή.